Ε, okay, we start this meeting, although... Λοιπόν, ξεκινάμε παρά το ότι δεν έχει έρθει ακόμα κανένας ε, βουλευτής, αλλά εμείς ακολουθούμε το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Ναι, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διερμηνία έχουμε. Σημείο 3, έγκριση των πρακτικών της 26 Σεπτεμβρίου. Συμφωνείτε, ναι. Και... Yes. Ε, ε, Τα, ξεκινάμε με το σημείο 4. Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης για την έκθεση της πρωτοβουλίας ΕΚΟΝ. Έχει αναβληθεί πολλές φορές. Και τώρα έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε και εκ παραλλήλου και θα κάνουμε και μια έκθεση για την νομοθετική έκθεση για την επέκταση του ΕΦΣΙΝ. Θα δώσω λοιπόν τον λόγο στην κυρία Ρωμάνα Τόμτς, την εισηγητρία. Έχετε τον λόγο. Hvala, hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Vsem seveda, ki ste tukaj in ste uspeli priti pravočasno, prav lepo dobro jutro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 I'm so sorry, I don't see Slovenian translator in... Do we have a problem with the interpretation? Έχουμε πρόβλημα με τη διερμηνία. It's box, it's box 20 for Slovenian inter... Δυστυχώς δεν υπάρχει διερμηνία από σλοβενικά Τουλάχιστον προβλεπόταν αρχικά, αλλά δεν βλέπω τους διερμηνείς. we don't Όχι, όχι, δυστυχώς δεν προβλέπονται σλοβενικά. Δυστυχώς. Θα προσπαθήσω να σας τα πω αγγλικά καταρχήν και θα, δεν θα μιλήσω όσο θα ήθελα. Νομίζω ότι θα δούμε το θέμα της διαρμηνίας αργότερα. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν είχα προετοιμάσει την ομιλία μου στα αγγλικά και ε, θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ, θα τα πω κάπως απ' έξω. Είχαμε λοιπόν πολλές ε, πολλά ζητήματα ως προς την έκθεση αυτή. Τώρα βρίσκεται επιτάπητος. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συνεργαστούμε και ελπίζω ότι οι σκιώδεις θα συνεργαστούν μαζί μου ο Κατάινεν, ο οποίος είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του ΕΦΣΙ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων μας ε, έχει πει ότι μας δίνει καλά αποτελέσματα. Αλλά δεν άκουσα καθόλου πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν χάρη στο Όπως αναφέρθηκε και πριν, ο βασικός στόχος των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από το ΕΦΣΥ είναι ακριβώς η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και να προκληθεί να δημιουργηθεί οικονομική ανάπτυξη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για τις ΜΜΕ, γιατί οι ΜΜΕ πραγματικά δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και επίσης θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις μικρότερες χώρες, διότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ΕΦΣΙ χρησιμοποιείται περισσότερο στις ε, χώρες, στις μεγάλες χώρες και έχουν επενδυτικά σχέδια και επενδυτικά προγράμματα που εντάσσονται στον εθνικό προϋπολογισμό. Όμως οι μικρότερες χώρες χρειάζονται περισσότερα χρήματα και θα πρέπει να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να εφαρμοστεί στις μικρότερες χώρες, να υπάρχει εύκολη, ευκολότερη προσβασιμότητα για τις μικρές χώρες. Το ΕΦΣΙ είναι ένα πολύ σημαντικό μέσον και έχει σημασία να επενδύσουμε στις κτηριακές εγκαταστάσεις, γέφυρες, σιδηροδρομικές συνδέσεις και ούτω καθεξής, αλλά φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι σήμερα έχει μεγάλη, μεγαλύτερη σημασία να επενδύουμε στους ανθρώπους, στο ανθρώπινο δυναμικό. Περί αυτού πρόκειται. Θα ήθελα λοιπόν να φτάσω στο συμπέρασμα ότι ελπίζω αυτή να είναι η αρχή της συνεργασίας μας και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα επανέλθουμε σε αυτά τα ζητήματα και ελπίζω ότι οι σκιώδεις θα συνεργαστούν και θα μπορέσουμε να συντάξουμε μια πολύ καλή έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορέσαμε να σας κατανοήσουμε πολύ καλά όλοι. Η, η Ιούτα έχει το λόγο που εκπροσωπεί τους σοσιαλδημοκράτες. Η Μιλιαν Πάβελ ε, απουσιάζει και μου ζήτησε να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει. Προσωπικά συμφωνώ με πολλά από αυτά τα οποία μόλις ε, μας είπατε. Ο κύριος Πάβελ θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων μπορεί να είναι ένα καλό μέσο για να δημιουργήσουμε την ανάπτυξη, να καταπολεμήσουμε την ανεργία και να απελευθερωθούν οι επενδύσεις στην Ευρώπη. Επίσης, θεωρεί ότι οι μικρόμεσες επιχειρήσεις στην Ευρώπη πρέπει να έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο. Τα έργα που θα χρηματοδοτούνται από το ΕΦΣΥ θα πρέπει να δημιουργούν θέσεις εργασίας καλές και βιώσιμες. Έχουμε εδώ πέρα ως στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών συστημάτων. ο Πάβελ συμφωνεί με την εισηγήτρια ότι η Κομισιόν αμέλησε την αξιολόγησή της να πει πόσες θέσεις εργασίας δημιούργησε το ΕΦΣΙ και σας ευχαριστεί και αναμένει τη συνεργασία με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Κύριο κύριος Κάλβε Σομπόν, αλλά δεν είναι εδώ. Οπότε περνάμε στην κυρία Βερμέγιο. Ούτε αυτή είναι εδώ. Τέρι Ράγκε, ούτε αυτή είναι εδώ. Και η Λάρα Άγκια δεν είναι εδώ αυτή. Να με άρεσε τον κύριο Μαρτίνα από το ΙΕΝΕΦ που είναι εδώ. <coughs> Euh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αρκετά γρήγορα φτάσαμε στο όνομά μου και εγώ. Θα ήθελα να πω τα εξή. Συμμεριζόμαι στα, στα γενικά τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένω και από την κυρία Εισηγήτρια Ε, που μας μίλησε προηγουμένως. Χαιρετίζουμε και τις ε, πρωτότυπες αυτές ιδέες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στατηγικών Επενδύσεων. Ξεκινάει με πολύ καλές προθέσεις, αλλά ξέρετε ότι θα υπάρξει ένα αλλά δημιουργία θέσεων εργασία, ε, μετάβαση στην βιώσιμη οικονομία, στήριξη προ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Πολύ καλέ προθέσει λοιπόν, αλλά είναι αδύνατο να αξιολογηθούν εφόσον οι μεταρρυθμίσει ε, συνεχίζονται για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ε, της ενισχυμένης ενιαίας αγοράς. Τα κακά αποτελέσματα... Χάνετε το μικρόφωνο του ομιλητή. Ε, δεν μπορούν να κρύψουν ε, τις ε, αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την, το διαθετικό πλαίσιο διαθετικών μεταρρυθμίσεων, μιας ε, σοβαρής και υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής και των επενδύσεων. Αυτό είναι που μας προβληματίζει γιατί θεωρούμε ότι αυτά τα ταμεία βασίζονται στην εφαρμογή από τα κάτι μελη διαθετικών μεταρρυθμίσεων. Και ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Ε, ιδίως οι χώρες που αντιμετωπίζουν ε, δυσκολίες. Αυτό σημαίνει μέτρα λιτότητας. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν πόρους μόνο όταν θα εφαρμόζουν αυτές τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις, δηλαδή μέτρα λιτότητας και αυτές τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις έχουν αποδείξει ε, ότι είναι αποτυχία. Δεν μπορούμε λοιπόν να στηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα σε καμία περίπτωση. Ευχαριστώ. Κύριε έχετε ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Ρωμάνα που με τα αγγλικά της μας έπεισε. Θεωρώ πως το ΕΦΣΙ είναι ένα ουσιαστικό μέσο με το οποίο μπορούμε να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Βεβαίω πρέπει και τα κράτη-μέλη να είναι διατεθειμένα να κάνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Εντάξει, είναι εύκολο να το λέει κανείς απ' έξω, αλλά υπάρχουν χώρες, όπως η Γερμανία, που έκαναν σοβαρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τώρα μπορούν να δουλέψουν, να επενδύσουν, να αλλάξει η κατάσταση. Και τα ποσοστά που έχουμε, ε, τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης, ε, χαμηλά ποσοστά ανεργίας δηλαδή, είναι ένδειξη του ότι αν κάποιος θέλει και έχει τη σύμφωνη γνώμη των κοινωνικών εταίρων μπορεί να καταφέρει πολλά. Πότε σημαντικό είναι αυτό το οποίο είπε Κομισιόν. Θέλουμε μια στρατηγική προσέγγιση να δώσουμε, να δώσει η Κομισιόν τη δυνατότητα να υπάρξουν τα σωστά αποτελέσματα. Η στόχη όμως πρέπει να είναι όχι να φτιάξουμε απλά κάτι δρόμους ή τίποτα γέφυρες, ή αυτό το οποίο είπαν κάποια κράτη-μέλη σε παλιά έργα. Α, ναι, ναι, ναι, αυτό να μα δώσει τώρα τα λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, δεν είναι αυτός ο στόχος. Εδώ έχει δίκιο η Ρωμάνα. Πρέπει να επενδύσουμε στους ανθρώπους. Έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να πούνε ναι, πρέπει να κάνετε κάτι. Να κάθετε και να περιμένετε να βρέξει λεφτά, δεν γίνεται αν κάνετε κάτι, ναι υπάρχουν λεφτά διαθέσιμα. Αν ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να δούμε τι γίνεται με τους νέους στην επαγγελματική απασχόληση. Να σου πούμε, ναι, για σας είναι κάτι θέμα να κάνουμε. Θεωρώ πως τότε θα έχουμε μια Ευρώπη η οποία θα έχει μια ουσιαστική προστιθέμενη αξία. κ. Ματέλη θα το κάνουν μόνο του τα κράτη-μέλη. Όχι, δεν το κάνουν. Δεν το έχουν κάνει. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πούμε πω είναι καλό να κινητοποιηθούν οι λογικές και οι σωστέ επενδύσεις. Έτσι ώστε τελικά ο κόσμος να νιώσει ότι είμαστε τμήμα μιας παραγωγικής εξέλιξης. Έτσι θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος από την Κομισιόν που θέλει να προσθέσει κάτι. Κύριε Χοκμάιρ, παραδείγματος χάρη. Όχι. Κάποιος άλλος, όχι. Η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Ας μιλήσει κάποιος. Πατάτε το κουμπάκι και μιλάτε. Εμεί ως Γενική Διεύθυνση Απασχόληση συμφωνούμε απολύτω ότι ε, αυτά τα άλλα στοιχεία και το ανθρώπινο κεφάλαιο θα πρέπει να αποφεληθούν ε, του ΕΦΣΥ. Σε αυτό το πλαίσιο συμμετέχουμε ενεργά προσπαθώντας ε, να συγκεντρώσουμε πόρους από διάφορα ενδιαφέρομενα μέρη προκειμένου να προάγουμε τα έργα του ΕΦΣΥ, τα οποία θα ε, δημιουργούν ε, περισσότερη και υψηλότερης ποιότητας απασχόληση με μεγαλύτερη κοινωνική αξία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Τόμς θέλει να επανέλθει συμπερασματικά. Εντάξει, δεν έχω και πολλά να πω, γιατί αρκετοί λείπουν σήμερα το πρωί. Ελπίζω αυτό να οφείλεται στην ώρα και όχι επειδή δεν μας ενδιαφέρει το θέμα. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ όλους όσοι ήρθαν ε, σήμερα το πρωί και σχολίασαν ε, τα όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και όπως είπα και προηγουμένως, ε, ευελπιστώ τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά στο μέλλον και ότι θα υπάρξει καλή συνεργασία με τους ε, σκιώδεις ε, εισηγητές. Σας ευχαριστώ. Εν είδη σύνοψης θα μπορούσα να πω ότι το ΕΦΣΥ, και αυτό είπαν κάποιοι από εσά. αξιοποιείται κατά κύριο λόγο από τις μεγάλες χώρες και μεγαλύτερες οικονομίες Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τα αποτελέσματα του ΕΦΣΕ. τουλάχιστον όχι σε αυτή τη φάση. Πόσες θέσεις απασχόλησης ε, δημιούργησε. Και κάποιοι από εσάς αναφέρατε ότι θα πρέπει να στηρίξουμε ή να θα πρέπει να στηρίξουμε αυτούς που εργάζονται, όχι αόρατες επενδύσεις ε, που κάπως να συνδέονται με την απασχόληση. Δεν είναι αυτός ο σκοπός του ΕΦΣΥ. Μεγαλύτερη απασχολησιμότητα λοιπόν. Και νομίζω ότι θα έχουμε την δυνατότητα να επανέλθουμε στη συζήτηση αυτή. Κρίμα που δεν είμαστε περισσότεροι σήμερα το πρωί, αλλά σας διαβεβαιώ ότι θα επανέλθουμε. Προθεσμή υποβολή τροπολογιών, η 6 Δεκεμβρίου και στην Επιτροπή μας ε, θα ψηφιστεί στις 25 ή 26 Ιανουαρίου. Και στην ε, Ολομέλεια θα τεθεί στη συνέχεια, να γνωρίζουμε ακριβώς πότε. Το επόμενο σημείο θα ξεκινήσει σε 9.45. Ο κύριος Πυρίνσκι που είναι εισηγητής δεν είναι ακόμα εδώ. Και εφόσον πρόκειται για τη συμφωνία ΣΕΤΑ, καλό είναι να περιμένουμε μέχρι την άφηξη του κύριου Πυρίνσκι. Θα κάνουμε λοιπόν ένα μικρό διάλειμμα. Δεν ξέρω τι θα πει τώρα. Α, δεν ξέρω τι θα πει τώρα. είναι πολύ ωραία. Να σας ενημερώσω ότι υπάρχει κίνηση, γι' αυτό καθυστερούν όλοι. Αλλά ελπίζω ότι σε μερικά λεπτά θα είμαστε έτοιμοι.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 στην ε, συνεδρία των Πρόεδρων των Επιτροπών εγώ επιχειρηματολόγησα για το δικαίωμα της Επιτροπής μας να έχει λόγο επί του θέματος και λήφθη μια απόφαση την ίδια μέρα στο Στρασβούργο και αυτό σημαίνει ότι ε, έχουμε την ευκαιρία τώρα και ο κύριος Πυρίνσκι σε ελάχιστο χρόνο κατάφερε να προετοιμάσει ένα σχέδιο γνωμοδότησης παρά το ότι ο χρόνος ήταν πολύ περιορισμένος. Θα του δώσω τώρα τον λόγο. Καθώς είναι ο εισηγητής για την θέση της επιτροπής μας στην ΣΕΤΑ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, Οπωσδήποτε το ζήτημα αυτό ήταν στο κέντρο των συζητήσεων τους τελευταίους μήνες, ίσως και χρόνια και θεωρώ ότι η Επιτροπή Απασχόλησης πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα γιατί είμαι πεπισμένος ότι η συμφωνία αυτή έχει άμεσες επιπτώσεις ακριβώς στα ζητήματα αρμοδιότητας της Επιτροπής μας. Απασχόληση, ανάπτυξη κτλ. Θα παρουσιάσω πολύ σύντομα λοιπόν το σχέδιο έκθεσης και τρία πράγματα θα προσπαθήσω να πω. Πρώτον, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι αναμφισβήτητα όσον αφορά την ΣΕΝΤΑ, τα οποία δεν α, ε, αμφισβητούνται. Πέντε από αυτά. Το πρώτο είναι ότι ε, δεν πρόκειται για μια απλή εμπορική συμφωνία. Το όνομα και μόνο λέει ότι είναι μια συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία. Δεύτερον, έχει αναγνωστεί ότι είναι μια μεικτή συμφωνία μεικτή αρμοδιότητα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν και των κρατών μελών. Και αυτό βεβαίω σχετίζεται με το ότι αφορά και τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου και όχι μόνο τις άμεσες επενδύσεις. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι η πρώτη συμφωνία του είδους της που κλείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια βιομηχανοποιημένη χώρα. Και κάποιοι την έχουν ονομάσει την πιο φιλόδοξη συμφωνία που έχει συναυθεί ποτέ από την Ένωση. Το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι η πρώτη συμφωνία με ένα λεπτομερές σύστημα επίλυσης διαφορών όπως λεγόταν και τώρα λέγεται ε, σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων. Προφανώς έχει πολλές και διαφορετικές επιπτώσεις και είναι ένα από τα πιο πολύ συζητημένα χαρακτηριστικά, αλλά είναι το, η πρώτη συμφωνία. Αυτό είναι το γεγονό. Και τέλο, οπωσδήποτε όχι είναι ότι είναι η πρώτη συμφωνία όπου στην σφαίρα των υπηρεσιών έχει εγκριθεί η αρνητική λίστα, όπως λέγεται. Δηλαδή η πρόσβαση στην αγορά για υπηρεσίες με βάση μια αρνητική λίστα πραγμάτων που αποκλείονται. Δεδομένων λοιπόν όλων αυτών των χαρακτηριστικών είναι σαφές ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή και λεπτομερής συζήτηση για το τι σημαίνει αυτή η συμφωνία η πρώτη του είδους της. Και εδώ πέρα δίνω τον λόγο στα στις τροπολογίες μου που αφορούν έξι η μία έχει να κάνει με τις θέσεις εργασίας και εδώ πέρα τα στοιχεία βεβαίω. δεν μας λένε αν θα έχουμε ακριβώς την δημιουργία θέσεων εργασίας που μας υπόσχονται. Μάλιστα το έγγραφο αυτό, την καλύτερη περίπτωση, μιλάει για την στήριξη, την διατήρηση θέσεων εργασίας. Αλλά αποφεύγεται τώρα να μιλήσουμε για δημιουργία. Οι μελέτες που έχουν γίνει μιλάνε για μια οριακή αύξηση και η μελέτη μιλάει για την απώλεια 200.000 θέσεων εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 10.000 στον Καναδά. Και βεβαίω η ανάλυση του Ιουνίου 2011 μιλάει ακριβώς για τα προβλήματα στο τομέα της απασχόλησης. Δεύτερον, η μισθή. Η έρευνα εδώ δείχνει ότι μάλλον θα υπάρξει μια αύξηση στο κενό εισοδήματος μεταξύ ειδικευμένων και μη ε, εργαζομένων ε, και η ανισοκατανομή ε, του πλούτου που θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη ανισότητα. Το τρίτο, έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εδώ πέρα και πάλι αυτοί που είναι υπέρ της συμφωνίας λένε ότι αυτό θα ωφελήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όμως και πάλι μόνο το 3% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ένωση εμπορεύονται με κόσμο εκτό της Ένωση ε, και το ίδιο ισχύει βεβαίω και με τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Τέταρτον, προστασία των εργαζομένων και αυτό έχει αναφερθεί. Υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ προστασίας των δικαιωμάτων και των εργαζομένων και της ε, διαδικασίας αυτής της συμβουλευτική που υπάρχει εδώ. Το επόμενο βεβαίω έχει να κάνει με το ότι θα υπάρξει μια διοχέτευση του εμπορίου που θα φύγει μακριά από τις χώρες και θα κατευθυνθεί πάλι σε μια βόρεια χώρα το οποίο πάλι θα δημιουργήσει προβλήματα μεταξύ αναπτυσσομένων και ανεπτυγμένων χωρών και έκτον των βεβαίως η νομική αβεβαιότητα υπάρχει ακόμα για το σύστημα των επενδυτικών δικαστηρίων. Ναι, βεβαίω. Υπάρχει. Το θέμα βέβαια στο οποίο δεν μας απασχολεί τόσο, γιατί και οι δύο χώρες έχουν ανεξάρτητα, και οι δύο πλευρές έχουν ανεξάρτητα συστήματα δικαιοσύνης και βεβαίω το επόμενο θέμα μας αφορά ιδιαίτερα ως κοινοβούλιο, ως ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο είναι η εμπιστοσύνη, η εμπιστοσύνη των πολιτών στους εκπροσώπους τους και στα θεσμικά όργανα που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους. Εδώ πέρα υπάρχει ένα έλλειμμα για να μποκρίσει εμπιστοσύνης και η όλη διαδικασία και τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία δύο χρόνια όταν οι διαπραγματεύσεις ε, ολοκληρώθηκαν κάπως απότομα. Δεν νομίζω πως έχουν προωθήσει και πολύ την εμπιστοσύνη στην διαδικασία. Δεν θα επέκταθω περισσότερο, ίσως μια άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you, Mr. Then we'll go to... Ευχαριστούμε κύριε Πυρίνσκι. Θα δούμε τώρα τους ε, σκιώδεις, τη θέση των σκιωδών. Η κυρία Τόντς από το ΕΛΚΑ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εμείς στο ΕΛΚ θεωρούμε ότι το ΣΕΤΑ είναι μια πολύ σύγχρονη και καλή συμφωνία, δίνει νέες ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα της ΜΜΕ και θεωρούμε ότι η ΣΕΤΑ προωθεί και διατηρεί υψηλές προδιαγραφές και θα μας ε, εγγυηθεί νέες θέσεις εργασίας. Έχει αυστηρούς νόμους για την προστασία του, των εργατικών δικαιωμάτων και του εργασιακού πλαισίου και καθίσταται σαφές ότι το ΕΛΚ δεν μπορεί να υποστηρίξει την πρόταση του εισηγητή. Ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να συνενέσει σε αυτή την πρόταση το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Η κυρία Τραβέσιους δεν ε, είναι παρούσα από το ECR. Ο κύριος Καλβέ Σαμπον και αυτός λείπει. Α, όχι, όχι. φτάσατε μόλις τώρα, έχετε το λόγο. Ε, προσπαθώ να τα καταφέρω ως προς τη φυσική μου ε, κατάσταση, αλλά όπως βλέπετε αυτό μπορεί ή μπορεί να μην έχει αντίκρισμα. Λοιπόν, θα συνεχίσω στα ισπανικά. Από πλευράς των ε, φιλελευθέρων, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν ε, ε, ορισμένες μικροαποχρώσεις σε σχέση με την έκθεση του εισηγητή. Και θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μία διαφορά 180 μοιρών από τη θέση του εισηγητή και τη δική μας. Θεωρούμε ότι μία συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ε, δημιουργεί θέσεις εργασίας, ε, οδηγεί σε αύξηση μισθών και ούτω καθεξής. Ε, δηλαδή, προσπαθούμε να αρθεί ο προστατευτισμός, αλλά υπάρχουν και στρατηγικοί για να εξασφαλίσουμε την ειρήνη, η οποία αποτελεί κοινωνικό αγαθό. Με τη σειρά της επίσης υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι ε, στόχοι ανανέωσης του παραγωγικού ιστού. Και αυτό αποτελεί προστιθέμενη αξία τη στιγμή που διαθέτουν και μεγαλύτερα, υψηλότερα μάλλον προσόντα. Άρα, για την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού αυτό αποτελεί ευεργέτημα. Και Μπορεί κανείς να βρει δουλειά σε τομείς που τον ικανοποιούν. Μπορούμε να ακολουθήσουμε το διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο ε, όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων. Δεν υπάρχει δηλαδή μία απλή ποσοστοποίηση ε, κερδών και θέσεων εργασίας. Αλλά θα ήταν παγίδα να σταθούμε μόνο σε αυτό. Εδώ αναφερόμαστε σε ένα κείμενο του 2011 όταν ε, διανύαμε τη μεγάλη οικονομική κρίση σε συγκυριακό επίπεδο, όπου έπρεπε να ληφθούν υπόψη πολλές μεταβλητές. Δηλαδή, μία συμφωνία ελευθέρου εμπορίου έχει σχέση με μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, δηλαδή σε 5, 10, 15 έως και 50 χρόνια. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ένας φωτεινός σηματοδότης με πόρτες ανοιχτές προς τον κόσμο. Δεν θέλουμε να σταθούμε στον προστατευτισμό. Γι' αυτό δεν ε, μας βρίσκει σύμφωνος το πνεύμα σύνταξης της έκθεσης. Φυσικά όλα τα πράγματα θα πρέπει να γίνονται όπως πρέπει και να μην υπάρχει μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με οποιοδήποτε κόστος και η τεχνολογική καινοτομία έχει επιπτώσεις στην εργασία. Θα την σταματήσουμε, όχι φυσικά. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και βραχυχρόνια, δηλαδή ως προς την ε, μεταβατική περίοδο που μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες. Αυτό θα πρέπει να το λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει πώς μπορεί να προστατεύσει και να βοηθήσει και αυτό εντάσσεται και στην συνολική συμφωνία ΣΕΤΑ. Θα μπορούσαμε λοιπόν στο κείμενό μας να υποστηρίξουμε την ιδέα ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις αρνητικές συνέπειες σε τομεακό επίπεδο, να προλάβουμε και ούτω καθεξής. Το Ταμείο για την Αντιμετώπιση της Παγκοσμιοποίησης μπορεί να συμβάλλει. Αλλά το να πούμε ότι η συμφωνία ε, με μια στρατηγική περιφέρεια του κόσμου που που αφορά ε, μια συμφωνία μεταξύ 35 εκατομμυρίων και 500 εκατομμυρίων από την άλλη πλευρά, ε, δεν είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει, το να λέμε ότι δεν θα δημιουργήσει θέσεις ε, εργασίας σίγουρα και δεν θα βοηθήσει την κατάσταση, δεν είναι μια αλληλέγγυα στάση, ούτε και θετική μέσα στα πλαίσια της ε, γεωστρατηγικής μας θέσης περί ειρήνης. Θεωρώ ότι ο προστατευτισμός ε, μας έδειξε τα αποτελέσματά του ιστορικά και γι' αυτό θα πρέπει να μην δεχτούμε αυτή τη θέση του εισηγήτη και θα υποβάλουμε τροπολογίες που αντιτίθενται σε αυτό το πνεύμα προστατευτισμού. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, η Τάνια Γκονσάλες Πένιας που εκπροσωπεί την ε, ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζουμε πολύ καλά τη ρητορική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς ε, και την ε, δημιουργία θέσεων εργασίας. Αλλά η ΣΕΤΑ δυστυχώς κατέρευσε στο κεφάλαιο 23 σε σχέση με το εργατικό δίκαιο. Σύμφωνα με μία μελέτη του Πανεπιστημίου ΤΑΦ στην ε, στο, στη ΣΥΠΑ, βλέπουμε ότι θα, υπάρχουν, θα υπάρχει μείωση εργασίας και θα χαθούν 250 θέσεις εργασίας. Θα υπάρχει μεγαλύτερη ε, απορρίθμιση, κάτι το οποίο δημιουργεί ανεργία και ευαλωτότητα στον τομέα της ενεργείας. Υπάρχει λοιπόν μια μεγαλύτερη πίεση των διεθνών αγορών που μειώνουν τις τιμές. Ο Καναδάς δεν δέχτηκε πολλές, ε, ε, πολλούς κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με μία συμφωνία ελευθέρου εμπορίου που θα οδηγήσει στην μείωση θέσεων εργασίας και πολλές απολύσεις και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 23 όπου υπάρχουν ε, εξαιρέσεις σε σχέση με διαδικασίες διαιτησίας. Δηλαδή η ΣΕΤΑ τι κάνει, ζητά από τα συμβαλόμενα μέρη να συμβάλλουν στην επίλυση των διαφόρων. Το κεφάλαιο 23.3.1 μιλά για επενδυτικά σχέδια, αλλά δεν υπάρχουν κυρώσεις εάν ένα κράτος μέλος ή ο Καναδάς ή οποιαδήποτε επιχείρηση παραβιάσει αυτό το πλαίσιο. Καθίσταται σαφές ότι και οι ξένοι απένδυτες θα πρέπει να προσφύγουν στα δικαστήρια εάν υπάρχουν επιπτώσεις επί των μισθών. Αλλά ε, δεν μπορούμε να δεχτούμε τους κανόνες της ΕΤΑ που πλήττουν τον κοινωνικό ιστό, γιατί και στην πνευματική ιδιοκτησία μπορεί να φτάσουμε σε αύξηση των τιμών, ακόμα και των ε, γενοσύμων. Και αυτό που έχει σημασία είναι να μην έχουμε μαζικές απολύσεις. Η ΣΕΤΑ ε, δεν απαγορεύει τους ε, φορολογικούς παραδείσους και δεν δημιουργεί αξιοπρεπή εργασία. Οι συλλογικές συμβάσεις και οι δημόσιοι διαγωνισμοί είναι αρκετά ευάλωτη και ε, δεν υπάρχει η ευεργεσία και η εγγύηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η ΣΕΤΑ μιλά για ε, δύο συναριακές ε, συμφωνίες δημοσίου συμφέροντος, αλλά στο κεφάλαιο των κεφαλαίων και υπηρεσιών ε, δεν εγγυάται την εργασία στη δημόσια υγεία και στα νοσοκομεία. Οι συμφωνίες σαν το TTIP και τη ΣΕΤΑ θα πλήξουν την Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία με υψηλούς δείκτες ανεργίας, ιδιαίτερα για τους νέους και με επισφαλή εργασία. Η ΣΕΤΑ δημιουργεί κινδύνους ως προς τα εργασιακά δικαιώματα και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να πλήξει την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Από τους ε, πρασίνους, την κυρία Ντελή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι ε, χαίρομαι που μπορώ να εκφράσω τη γνώμη μου σε αυτή την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. το θέμα της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς κάνουμε ένα βήμα μπρος, ε, δύο βήματα πίσω. Αυτό έχει κάνει ο κύριος Σούλς ε, και με, με τον μεγάλο συνασπισμό ε, το τελευταίο διάστημα. Αυτό έχει επιπτώσεις. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στην έκθεση της Επιτροπής μας πριν για αυτό το ζήτημα ενώ παράλληλα εξετάζουμε τέτοια ε, ζητήματα ευρύτερα των εργασιακών και στέκομαι σίγουρα ε, και ε, στον ρόλο των Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών για τη Δημοκρατία. Ευχαριστώ τον κύριο Βιρίνσκι για το περιεχόμενο του σχεδίου νομοδότησής του. αναδεικνύει πραγματικά τον πυρήνα του ζητήματος. Αυτές ε, οι υποσχέσεις ε, για άνοδο της κοινωνικής συνοχής και των εργασιακών συνθήκων στην Ευρώπη μπορώ να σας πω ότι πρόκειται για χήμερες αγαπητοί συνάδελφοι. Μας πουλάνε φύκη και μεταξυτές χορδέλες. Η πραγματικότητα είναι ότι ε, θα χάσουμε πράγματα. Αντί λοιπόν ε, να ε, προσπαθούμε να επιβάλλουμε πολιτικές, ας ακούσουμε λίγο με σεβασμό τους ε, πολίτες. Η ΣΕΤΑ δεν ανταποκρίνεται καθόλου στις σημερινές προκλήσεις. Ο φόβος των πολιτών τι είναι. Είναι ο αριθμός των 25 εκατομμυρίων ανέργων στην Ευρώπη. 25 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω. Είναι η ενεργεία σήμερα, όχι σε 20 χρόνια. Α είμαστε λοιπόν λίγο υπεύθυνοι αλλά και φιλόδοξοι πάνω απ' όλα. Εμείς στο νομοθετικό μας έργο θα πρέπει όντως να παρουσιάσουμε μια εναλλακτική λύση για να αντιμετωπίσουμε αυτή την αργία. Είναι πολύ απλή αυτή η εναλλακτική. Μια εναλλακτική που θα στέλνει που θα δείχνει το βαθμό στον οποίο είμαστε ε, σε θέση να αλλάζουμε την πραγματικότητα των πολιτών χάρη ακριβώ στην ενεργειακή μετάβαση στην ε, επανέναρξη της οικονομίας, της ε, επαναδιοχέτευσης των εργαζομένων σε άλλους ε, κλάδους. Ας πούμε εδώ αναφέρουμε στην αυτοκινητοβιομηχανία. Επομένω, πρώτα απ' όλα πρέπει να απορρίψουμε αυτή τη συμφωνία της ΣΕΤΑ. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε το σχέδιό σας, κύριε Σιγητά, και ελπίζουμε ότι αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης θα τύχει ευρεία στήριξη στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε δεν είναι εδώ. Τι να ο κύριος Μαρτέν, τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πάλι παραδόξως συμμεριζόμαστε το σκεπτικισμό του κυρίου Πυρίνσχη. Μάλιστα συμφωνούμε μαζί του. Πράγματι, στην ε, αιτιολογική του έκθεση μας ε, εξηγεί, συγγνώμη που επαναλαμβάνω τα όσα λέτε, αλλά συμφωνώ απολύτως. Μας εξηγεί λοιπόν ότι παρότι οι τελικές συνέπειες της ΕΤΑ είναι η ε, αύξηση της απασχόλησης, η ισορροπημένη μισθή και επιχειρηματικότητα, τα εμπειρικά δεδομένα που προκύπτουν από πραγματικά μοντέλα μας δείχνουν ε, οριακές αυξήσεις ε, συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ξεπερνούν το 0,018% σε μια περίοδο 6 έως 10 ετών εφαρμογής της συμφωνίας. Ο κύριος Πυρίνσκι επίσης αναφέρει ότι ε, οι προβλέψεις μιλούν για μείωση των θέσεων εργασίας μερικών χιλιάδων θέσεων ε, απασχόλησης, 45.000 στη Γαλλία, 42.000 για την Ιταλία, 19.000 ε, για τη Γερμανία. Και προβλέπεται και αύξηση της ανεργίας. Σε ό,τι αφορά τους μισθούς, τα στοιχεία δείχνουν ότι η συμφωνία θα διεύρυνε το χάσμα ε, μεταξύ των ε, ε, ανειδίκευτων εργατών και των ειδικευμένων. Και έτσι αυξάνονται και οι ανισότητες και οι κοινωνικές εντάσεις. Έτσι αναφέρει ο εισηγητής. Η συμφωνία δεν συμπεριλαμβάνει κανένα κεφάλαιο για συγκεκριμένα μέτρα στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 20,9 εκατομμύρια τέτοιες επιχειρήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση Μόλις 600 κάτι χιλιάδες όμως εξάγουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε έναν απελευθερωμένο περιβάλλον ε, της ΣΕΤΑ, αυτές οι μικρές επιχειρήσεις ε, θα εκτεθούν ε, σε έναν απίστευτο ανταγωνισμό των πολυεθνικών της, της Βόρειας Αμερικής και έτσι τίθενται σε κίνδυνο 90 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη διαφορά μεταξύ του επίπεδου ε, προβλεπόμενης ε, προστασίας για τους επενδυτές, για τα συμφέροντα και για τα εργασιακά δικαιώματα. Όλα αυτά έρχονται σε μεγάλη αντίθεση με τον μηχανισμό ε, διαβούλευσης που προβλέπεται για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Από πλευρά εξηγήσεών του, λοιπόν, ο κύριος Πυρίνσκι ενθαρρύνει την Επιτροπή ΙΝΤΑ, που είναι καθήλυνα αρμόδια, να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην δώσει τη συγκατάθεσή του για τη ΣΕΤΑ. Είναι πολύ σαφής, θέλει να μην εγκρίνει τη ΣΕΤΑ. Και έχω την εντύπωση ότι θα σας ε, στηρίξουν ε, από ό,τι έχω ακούσει από τους επιμέρους ομιλητές. Κύριε Πυρίνσκι, αν διατηρήσετε τη θέση σας, είναι σαφές ότι και εμείς θα σας στηρίξουμε, γιατί για εμάς η ΣΕΤΑ είναι προφανές ότι είναι στο ίδιο μήκος κύματος με την TTIP ή με την ΤΑΦΤΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αρένα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Έχω την ευκαιρία να είμαι ταυτόχρονα και στην ΙΝΤΑ ε, και εδώ πληρωματικό μέλο στην Επιτροπή Απασχόληση και χαίρομαι γιατί υπάρχει γνωμοδότηση ε, τη Επιτροπή Απασχόληση για ακριβώ αυτό το ζήτημα. Όπω θεωρώ ότι θα υπάρχει τέτοια γνωμοδότηση για όλε τι εμπορικέ συμφωνίε που εξετάζει η ΙΝΤΑ. Γιατί ε, η πλειονότητα των μελετών ε, στις οποίες αναφέρεται ο κύριος Πυρίνσκι δείχνουν ότι η πρώτη επίπτωση αυτών των εμπορικών συμφωνιών αφορά ακριβώς τα εργασιακά. Απασχόληση, δημιουργία θέσεων απασχόλησης ή όχι, ή ακόμα και απώλεια θέσεων απασχόλησης, αλλά και αντίκτυπος ε, στους μισθούς, ε, στην μετατόπιση των θέσεων εργασίας. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν και νικητές, αλλά υπάρχουν και χαμένοι και ξεκινούμε από την υπόθεση ότι αυτοί οι χαμένοι μπορούν να κινηθούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μεταφέρουμε εύκολα έναν Σουηδό εργαζόμενο προς την Νότια Ιταλία. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν μεταφέρεται τόσο εύκολα ένας ε, Ρουμάνος αγρότης για να γίνει ένας εργαζόμενος ε, των νέων τεχνολογιών στη Γερμανία. Δεν είναι τόσο εύκολα αυτά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να τα λάβουμε υπόψη όλα αυτά στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που εξετάζουμε στην ΙΝΤΑ. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει και αυτή η γνωμοδότηση. Θα απαντήσω στον κύριο Τσαμπών σε αυτά που είπε. Είπε ότι με τους Καναδούς συμμεριζόμαστε τις ίδιες αξίες. Σύμφωνα αρκετά μαζί του. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε τις καναδικές ε, ε, αξίες για να πούμε πρέπει να στηρίξουμε αυτή την πρόταση γιατί έχουμε τις ίδιες αξίες. Όταν μιλούσαμε για την συμφωνία με, τις, ε, με τους Αμερικανούς λέγαμε δεν έχουμε τις ίδιες αξίες αλλά πρέπει να την κάνουμε τη συμφωνία. Όταν μιλούμε για συγκεκριμένε αφρικανικέ χώρε και μάλιστα δικτατορίε, πάμε με κλειστά τα μάτια. Τι ξεχνάμε τι αξίε ξαφνικά. Εξετάζουμε λοιπόν στην ίντα τη διευκόλυνση εμπορίου με την Τουρκία, ενώ μόλι στο Κοινοβούλιο ψηφίσαμε ότι θα πρέπει να παγώσουν οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία εξαιτία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ είμαι η πρώτη που λέει ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για τις αξίες. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να αλλάζει ανάλογα με τις ε, συμφωνίες. Αν είναι να μιλήσουμε για αξίες θα μιλάμε για πάντα. Και όχι όταν μας συμφέρει μόνο. Είναι σημαντικό αυτό. Επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Πυρίνσκι. Η ανάπτυξη 0,23% ε, μέσα στη δεκαετία, στην καλύτερη περίπτωση. Από την άλλη, ε, βλέπουμε από όλες τις μελέτες ότι αυτό έχει επίπτωση ε, στις θέσεις απασχόλησης και στην κινητικότητα. Αν πάρουμε, για παράδειγμα, τους αγρότες, αυξάνοντας τις εξαγωγές ποσοστώσεων χείριου και βόηου ε, κρέατος υπάρχουν κλάδοι της οικονομίας που θα πληγούν, δύσκολα θα ανακτήσουμε αυτές τις θέσεις απασχόλησης. Για τους μισθούς οι χαμηλοί μισθοί θα χάσουν ε, περισσότερο. Υπάρχει όντω αύξηση στου υψηλού μισθού, όμω αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται, εντείνονται οι αντιθέσει στην Ευρώπη. Επομένω, αντί να πούμε α ψηφίσουμε τη ΣΕΤΑ και μετά βλέπουμε, εγώ θα έλεγα αντίθετα να τα εξετάσουμε. Να προβλέψουμε και να ε, θέσουμε σε ισχύ οτιδήποτε θα χρειαζόταν για να προσαρμόσουμε την ε, οικονομία μας και την κοινωνία μας σε ένα τέτοιο πλαίσιο και μετά να την υπερψηφίσουμε. Όχι να τα κάνουμε ανάποδα τα πράγματα. Να θέσουμε σε εφαρμογή οτιδήποτε θα μπορούσε να προβλέψει και να, να αποφύγει τέτοιου είδους ε, θέσεις απασχόλησης πριν ψηφίσουμε τη ΣΕΤΑ. Κύριε Μπάλλας, θέλετε το λόγο ή για το επόμενο θέμα. Παρακαλώ. Non, je vais être rapide puisque l'essentiel des... Πολύ σύντομα, γιατί οι συνάδελφοι ήδη Πυρίνσκι και τώρα η κυρία Μαρία Ρένα μόλις ανέφεραν τα, τα σχόλια που ήθελα να κάνω κι εγώ. Ήθελα μόνο να κάνω ορισμένες επισημάνσεις. Πολύ συχνά αναφέρεται ότι η αριστερά, οι προοδευτικοί ε, τυφλώνονται από την ιδεολογία και ότι δεν είναι συνεπείς και ρεαλιστές. Θέλω να αντιστρέψω αυτή την ψευδή φήμη Νομίζω ότι ο κύριος Πυρίνσκι έχει κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια, να πάει σε βάθος και να εξετάσει ενδελεχώς αυτές τις μελέτες. Πρώτη διαπίστωση, είναι σπάνιες αυτές οι μελέτες. Ε, για κάποιους είναι οι μελέτες του 2011 της Επιτροπής, ε, κάποιες είναι έξω ευρωπαϊκές, αναφέρεται. Και αυτό που είπε η κυρία Ρένα για την αυστριακή ε, μελέτη είναι ότι στην καλύτερη περίπτωση έχουν ε, διαφορετικά συμπεράσματα ή μπορεί να είναι και ιδιαίτερα απεσιόδοξες για τις ε, επιπτώσεις ε, της ΣΕΤΑ. Εγώ θέτω το ερώτημα. Γιατί θέλουμε να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία ΣΕΤΑ. Κανένα λογικό στοιχείο δεν μας λέει σήμερα ότι αυτό θα ωφελήσει όπως αναφέρεται στο, στην αιτιολόγηση της ΕΤΑ, δεν θα έχει λοιπόν θετικές επιπτώσεις στις ε, μικρότερες επιχειρήσεις, στην απασχόληση κτλ. Γιατί να το κάνουμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εγώ νομίζω ότι συνδέεται με την ιδεολογία. Δηλαδή, σήμερα έχουμε ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες που λένε ότι κατανοούν μια νέα ε, συμφωνία ε, και τις συνέπειες της μάλλον της ΕΤΑ, ε, ανησυχούν γιατί υπάρχει ένας προστατευτισμός και ότι θα επιστρέψουμε ουσιαστικά, θα κλείσουμε τα σύνορα, θα επιστρέψουμε στη δεκαετία του 30 και στον πόλεμο. Αυτό είναι ουσιαστικά. Και εγώ θέλω να φύγει αυτός ο εφιάλτης από ε, την πραγματικότητα. Εμείς έχουμε εμπορικές σχέσεις σήμερα και με τον Καναδά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ουσιαστικά σε ένα πλαίσιο ελευθέρων συναλλαγών, τουλάχιστον ως προς τα τελωνιακά. Βλέπουμε ότι αυτές οι νέες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που μας προτείνονται αυτή τη στιγμή δεν είναι παραδοσιακές ε, συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που αφορούν το εμπόριο δηλαδή, όμως ε, επιμένουν κυρίως σε μια αλλαγή προτύπων και νόμων και κυρίως σε ό,τι αφορά την ε, δυνατότητα προστασίας ιδιωτικών επενδύσεων με τον έναν τον άλλον τρόπο. Δεν θέλουμε λοιπόν να αυξήσουμε τις εμπορικές συναλλαγές για να αυξήσουμε την απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα. Θέλουμε να δώσουμε περισσότερη εξουσία σε ανθρώπους που ήδη την κατέχουν, που είναι πολυεθνικές. Δεν ξέρω αν η σκιώδης ε, του ΕΛΚ είναι εδώ, γιατί ήθελα να μας ακούσει, γιατί έχουμε αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε έναν διάλογο, που δεν θα το έχουμε για πολύ καιρό. Αλλά εξετάζουμε τα δεδομένα σήμερα για τη ΣΕΤΑ και στα στοιχεία, στα δεδομένα, τίποτα δεν μας δείχνει ότι θα ωφελήσει την Ευρώπη και τα λίγα πενιχρά στοιχεία που έχουμε μας δείχνουν ότι θα είναι μάλλον αρνητικές οι επιπτώσεις. Επομένως και με απόλυτα λογικό τρόπο πρέπει να, ακολουθήσουμε τη γνώμη του συναδέλφου Πυρίνσκι. Σας ευχαριστώ η κυρία Τόμτς έφυγε, αλλά ε, έκανε κάποιες παρατηρήσεις πιο πριν, οπότε περνάμε στον κύριο Λεπικάρτη, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάζοντας αυτό εδώ το έγγραφο και ακούγοντας τα σχόλια, να αν ζούμε στον ίδιο πλανήτη. Δηλαδή 37 κοινοβούλια έχουν συμφωνήσει πάνω σε αυτό το θέμα, οι κυβερνήσει σε όλο τον κόσμο. Αναμφισβήτητα θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ε, απασχόλησης ε, και για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Αναμφισβήτητα. Οπότε τι, τι κάνουμε σε αυτήν την Επιτροπή. Αναρωτιέμαι. Είναι παράλογο. Για να είμαι σαφής. Εμείς στην Άλντε στηρίζουμε με όλη μας την καρδιά τη συμφωνία αυτή. Και ευτυχώς, ευτυχώς και η μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Γιατί ακούγοντα συζήτηση αυτή σου γεννιούνται αμφιβολίες. Να προσθέσω λίγα σχόλια σε αυτά τα νούμερα που περιέχονται εδώ. Η μελέτη αυτή είναι ακόμα ένα έγγραφο εργασία. Δεν έχει μελετηθεί από άλλους επιστήμονες. Αυτό είναι γεγονό. Μία από τις βασικές τη ε, συνεισφορέ είναι ότι χρησιμοποιεί άλλο οικονομικό μοντέλο, διαφορετικό από αυτό το οποίο συνήθω χρησιμοποιείται στις αξιολογήσει αντικτύπου, γιατί δεν το λέει κανείς. Αν δείτε όλα όσα έχουν δημοσιευτεί μέχρι στιγμή. η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου έχει βγάλει ένα φύλλο με χρήσιμες πληροφορίε για τα οικονομικά ωφέλη της ΣΕΤΑ. Αν δείτε τον ΩΣΑ, στη δικιά του τη σελίδα, πολύ χρήσιμες πληροφορίε για τα εμπορικά ωφέλη και τα ωφέλη στην απασχόληση. Εδώ πέρα βλέπουμε μια ενδιαφέρουσα δήλωση. Και αναφέρω επιλέξη από τις 14 ε, ε, κύριες μελέτες που έχουν γίνει από το 2000 ε, που εξετάστηκαν και οι 14 και οι 14 συμπεραίνουν ότι το εμπόριο παίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση των εισοδημάτων. Και εμείς μιλάμε εδώ πέρα με με ένα έγγραφο εργασία και όχι με μελέτες ε, που έχουν εξεταστεί από άλλους επιστήμονε. Αν δούμε τα γεγονότα λοιπόν, αναφέρθηκε ότι η ΣΕΤΑ θα είναι η πρώτη συμφωνία με μια βιομηχανοποιημένη χώρα. Είναι γεγονός αυτό. Δηλαδή αν δούμε τη συμφωνία με την Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα είναι επιδημοκρατοποιημένη χώρα. Ας δούμε τα γεγονότα λοιπόν. Οι εξαγωγές της Ένωσης στην Νότια Κορέα αυξήθηκαν κατά 55% των απελευθερωμένων αγαθών κατά 57%. Οι εισαγωγές των πλήρως και μερικώς απελευθερωμένων προϊόντων αυξήθηκαν 35% ε, και 64% αντιστοίχως. Οπότε ε, λειτουργεί και για την Νότια Κορέα η συμφωνία. Οπότε το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε πλεόνασμα με την Νότια Κορέα. 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, ευρώ το 2015. Τελείως διαφορετική εικόνα δηλαδή. Ε, αν δείτε τα γεγονότα. Όπως είπα, η ομάδα της Άλτε στηρίζει πλήρως συμφωνία αυτή και ελπίζω η Επιτροπή μας να συνέλθει κάποια στιγμή. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε το κείμενο αυτό καθόλου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κέλλερ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αυτοί που είναι κατά της ε, ΣΕΤΑ συχνά παρουσιάζονται ως ε, κάποιοι που θέλουν να βλάψουν τον Καναδά. Γι' αυτό ζητήσαμε τη γνωμοδότηση διαφόρων καναδικών συνδικάτων και η θέση τους είναι αρνητική. Οι ίδιοι οι Καναδοί λένε ότι οι εκτιμήσεις ε, των όφελων είναι αμφισβητούμενες και αβεβαίες και ζητάνε κάποια προστασία του περιβάλλοντος ε, και των εργαζομένων που θα πηγαίνει πέρα από διακήρυξης ε, προθέσεων. Το δε νέο σύστημα αυτό επίλυση διαφορών δεν αλλάζει το ότι μόνο οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφεύγουν και οι κυβερνήσεις απλά να υπερασπίζονται αυτόν. Και ο Καναδάς αυτή τη στιγμή ε, είναι στα δικαστήρια με μεγάλες επιχειρήσεις για 8 δισεκατομμύρια δολάρια καναδικά. Οποιαδήποτε προσπάθεια να ρυθμιστούν στρατηγικοί τομείς είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για τις κυβερνήσεις γιατί οι κυβερνήσεις δεν ξέρουν πότε θα τους μηνύσουν κάποιες επιχειρήσεις. Οι ναι, παρουσίες ή οι μελλοντικές ε, υπηρεσίες δεν αναφέρονται στον κατάλογο υπηρεσιών προς απελευθέρωση. η ε, Γίναν δύο-τρεις ε, παρατηρήσεις από τον κύριο Στίγκλιτς, νομπελίστα, κατά της ΣΕΤΑ και δεν πρέπει να τον θεωρήσουμε ότι ούτε αυτός δεν καταλαβαίνει την οικονομία. Εμείς λέμε πως η Ευρώπη έχει την αλληλεγγύη ως μία αξία κλειδί. Συμφωνώ με αυτό και θεωρώ ότι το να είμαστε κατά της συμφωνίας αυτής είναι ακριβώς ε, επίδειξη αλληλεγγύης με τα καναδικά συνδικάτα και τους καναδούς πολίτες που είναι επίσης κατά αυτής της συμφωνίας. Ε, ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύτηκε 7 χρόνια με τον Καναδά κατόπιν εντολής των κατανολών. Τρεις ερωτήσεις έχω προς τον ε, κύριο Σιγητή. Είστε κατά όλων των εμπορικών συμφωνιών. Δεύτερον, δηλαδή, ε, αν δεν κάνουμε εμπόριο με τον Καναδά, με ποιον θα κάνουμε εμπόριο, το είπατε και μόνοι σας, έχουν τις ίδιες αξίες με εμά, επιμένουν στα κοινωνικά, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη δημοκρατία, στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα μπορούσα να συνεχίσω. Τρίτον, ασκήσατε κριτική στη διαδικασία, γιατί σε τα γνωρίζατε ότι τα κράτη-μέλη ενέκριναν ομόφωνα μία διαπραγματευτική εντολή και η Κομισιόν ακολούθησε πλήρω όλου αυτού του στόχου. Ε, πραγματικά δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω δηλαδή. Επί της αρχής είμαι αντίθετος με την θέση σας και συμφωνώ με του συναδέλφους μου στην ομάδα του ΕΛΚ. Οποιαδήποτε συμφωνία είναι καλύτερη από το μοσαϊκό που έχουμε τώρα. Ένα μοσαϊκό το οποίο δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα από την συμφωνία αυτή. Έστω και αν δεν είναι ιδεώδης για όλους μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φουντούλης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ΣΕΤΑ, όπως και η TTIP, είναι δύο όψεις του δύο νομίσματος. Δυστυχώς στην Ολομέλεια η πλειοψηφία ψήφισε να μην εισαχθεί η ΣΕΤΑ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για νομικό έλεγχο. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι αυτές οι εμπορικές συμφωνίες νέας γενιάς σκοπεύουν να μετασχηματίσουν το θεσμικό πλαίσιο προς όφελος των πολυεθνικών. Επίσης, αναφέρονται σε πολύ περισσότερου τομεί τη ζωή μα εκτό από το εμπόριο. Διαμορφώνεται ένα σύστημα διαιτησιών από ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία που θα επιτρέπει την αμφισβήτηση κάθε εθνική προστατευτική νομοθεσία, που θα περιόριζε τα κέρδη των πολυεθνικών εταιριών και θα άφηνε περιθώρια για μεγάλε οικονομικέ διεκδικήσει από αυτέ. Η συμφωνία αυτή βάζει το διεθνέ εμπόριο πάνω από τη δημοκρατία, τα κεκτημένα δικαιώματα των πολιτών, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και δίνει υπερεξουσίες σε επιχειρήσεις και πολυεθνικά λόμπι, ώστε να παρακάπτουν κυβερνήσεις και νομοθεσίες αν κρίνουν ότι θίγονται τα συμφέροντά τους. Όσον αφορά την Επιτροπή μας, τίποτα δεν μας εγγυάται την αύξηση των θέσεων απασχόλησης, αλλά οι εργαζόμενοι θα δουν τα δικαιώματά τους να περιστέλλονται περαιτέρω στο όνομα του κέρδους. Η αλήθεια είναι πως κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα τα ωφέλη. Σε πολλές περιπτώσεις, τέτοιου είδους οικονομικές συμφωνίες έχουν οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας, όπως για παράδειγμα με την περίπτωση της ναύτα μεταξύ ΙΠΑ, Καναδά και Μεξικού. Εάν η ΣΕΤΑ εφαρμοστεί, αλλά και η TTIP που έρχεται, θα προκαλέσουν την απώλεια περισσότερων από ενό εκατομμυρίου θέσεων εργασίας σε Καναδά, ΙΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. έχει το Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ορισμένα σχόλια και από τη ε, δική μου πλευρά συμφώνω με τον κύριο Σαμπών σε σχέση με αυτά που προανέφερε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να το δούμε και από πλευράς κοινωνικής και οικονομικής. Δηλαδή η Επιτροπή ε, απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων θα πρέπει να ασχολείται με δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Μιλάμε για κοινωνικά αγαθά που εντάσσονται σε μια κοινωνική πολιτική γενικότερα και αυτό μέσα στους γενικότερους ε, γεωστρατηγικούς στόχους. Αυτό είναι το πλαίσιο των συζητήσεων μας. Όταν οι πολίτες ρωτούν πώς θα ευεργετηθούμε από αυτή τη συμφωνία. Ένας, αν ένας άνθρωπος στο δρόμο σας, ζητούσε, σας ρωτούσε κάτι τέτοιο, δηλαδή ποιο είναι το τελικό ευεργέτημα, τι θα λέγαμε. Συμφωνώ με τον Ενρίκε. Δεν ξέρουμε αν θα δημιουργήσει περισσότερες ε, και θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι το ευεργέτημα είναι περιθωριακό. Αν δούμε και την ε, μελέτη αντικτύπου της Επιτροπής, γίνεται λόγος για 0,2% έως 0,5% πραγματική αύξηση του ΑΕΠ μακροχρόνια. Ε, αυτό δεν είναι μηδενικό δηλαδή, αλλά δεν είναι και σημαντικό. Και έγινε λόγος για τα πρότυπα που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, ένα υπολογιστικό πρόγραμμα το οποίο μιλά για δημιουργία πλήρους απασχόλησης. Ξέρουμε ότι αυτό είναι ανέφικτο, όπως είπε και η Μαρία Ρένα. Εάν ένας αγρότης στη Ρουμανία χάσει ε, οποιαδήποτε ε, πηγή εργασίας δεν είναι το ίδιο με κάποιον που θα χάσει την εργασία του στο Δουβλίνο ή στο Παρίσι. Δεν είναι αυτή η πραγματική ζωή. Ναι, ε, χάνονται και κερδίζονται θέσεις εργασίας, αλλά όταν μιλάμε για ένα πλαίσιο εγγυήσεων, εγγυήσεις έχουν μόνο οι επενδυτές. Κανένας άλλος και δεν κατανοώ πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να περάσει αυτό το μήνυμα. Δηλαδή ότι υπάρχει εγγύηση μόνο για τους επενδυτές και όχι, αυτό, και όχι στα ε, τακτικά δικαστήρια αλλά και, στα, ε, και σε εξειδικευμένα δικαστήρια, το ΔΕΚ γιατί λέμε στους εργαζόμενους ναι, μπορούμε να κερδίσουμε ε, θέσεις εργασίας, αλλά μπορείτε να χάσετε τη δική σας και δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε τίποτα. Και ε, μην ξεχνάμε ότι και το Ταμείο αντιμετώπισης της παγκοσμιοποίησης έχει χάσει τα δύο τρίτα των εσόδων του χωρίς εγγυήσει από την Επιτροπή ότι θα υπάρξει αύξηση κονδύλιων προς αυτό. Αυτό δεν είναι λύση λοιπόν. Τέλος πολλές φορές μιλάμε για το ε, πάγωμα που μπορεί να υπάρξει από πλευράς δικαστηρίου επίλυσης διαφορών. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ε, τι μας προτείνει η Επιτροπή. Τα κράτη έχουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν για ρύθμιση Δηλαδή δεν περιμένουμε έναν από Θεό να επιλύσει όλα μας τα ζητήματα, αλλά το ζήτημα είναι πώς μπορεί να συνεισφέρει για να επιλύσει μερικώς ορισμένα από τα ζητήματά μας. Δέχομαι το γεωπολιτικό χαρακτήρα, δέχομαι τις αξίες μας, δεν τις αγνοούμε, αλλά πού υπάρχουν ατράνταχτα στοιχεία για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δεν υπάρχουν. Ο συνάδελφος ο Μάρτι μίλησε για 27 ή 28 κράτη που το συζήτησαν και συμφώνησαν. Δεν ξέρω για τους άλλους συναδέλφους, αλλά στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο δεν έγινε καμία συζήτηση, καμία συζήτηση για αυτή τη συμφωνία. Έγινε ε, μία συζήτηση στη Γερουσία που την απέρριψε την απέρριψε η δική μας ανοβουλή. Δεν ξέρω λοιπόν τι έγινε στα άλλα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω κατά πόσο έγινε μία ευρεία σε εμβέλεια συζήτηση όπως θα έπρεπε να είχε γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κρίστινσεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν είχα σκοπό να λάβω το λόγο, γιατί δεν συμφωνώ με τους περισσότερους τους της ομάδας μου όταν λένε ότι οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου είναι κακές. Αλλά επειδή είμαι σοσιαλιστής και δημοκράτης, υποστηρίζω τις... Ε, ε, συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Δηλαδή η ΕΚΑΧ το 51 όταν ιδρύθηκε, ιδρύθηκε για αυτό το λόγο. Για να υπάρχει μία αλληλεγγύη. Και σήμερα οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση γι' αυτό. Δεν εστιάζουμε σωστά το θέμα μας. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συνάψει συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου ανά τον κόσμο, όπως ε, κάνουμε στην εσωτερική αγορά, αν δεν θέλουμε να το κάνουμε, τότε τι λόγο ύπαρξης έχουμε. Διότι είχαμε την οικονομική κρίση του 2008 και αυτό ε, ε, ε, οδήγησε σε μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας. Δηλαδή αφορούσε τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος κατέρευσε και κακοδιαχειρίστηκε ε, την, αγορά χρήματος, την αγορά κεφαρέων. Δηλαδή, οι δυνάμεις της αγοράς δεν μπορούν να μας καταδυναστεύουν. Εμείς θα πρέπει να τις ορίζουμε. Εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω μία συμφωνία ελευθέρου εμπορίου που δεν ε, προβάλλει συγκεκριμένες αξίες υπέρ των ε, εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά δεν μπορούμε να χτίσουμε τείχους και να απομονωθούμε από, τη, τον, επόμενο, από τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν κατανοώ αυτή τη συζήτηση. Κατανοώ ότι οι άνθρωποι δεν νιώθουν ασφαλείς γιατί είναι πολύ άνεργοι στην Ευρώπη αλλά εάν βάλουμε τροχοπέδες παντού, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ αυτή την προσέγγιση στο ελεύθερο εμπόριο. Ευχαριστώ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η οποία θα συνεχιστεί όταν θα φτάσει σύντομα η Επίτροπος Μάλστρομ. Να δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Πυρίνσκι Όπως είπα στην αρχή, υπήρχαν κάποιες επιτροπές που για πολύ περίεργους ε, λόγους δεν τους επιτράπει να γνωμοδοτήσουν για τη Συμφωνία ΣΕΤΑ. Και αποφασίστηκε για τη δική μας Επιτροπή Απασχόλησης και για την Επιτροπή Μεταφορών, για παράδειγμα, μόλις την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Ήταν πολύ περίεργο όλο αυτό. Γιατί όπως ε, ακούσαμε είναι εξαιρετικά σημαντική συζήτηση το θέμα του εμπορίου και οι συνέπειες που έχει το εμπόριο στην απασχόληση και στο κοινωνικό θεματολόγιο. Ο κύριος Πυρίνσκι είχε πολύ λίγο χρόνο στη διέθεσή του, αλλά τα κατάφερε. Παρακαλώ, κύριε Πυρίνσκι, αν έχετε μερικά καταληκτικά σχόλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση. που κατά πολλούς τρόπους δεν είναι η συνήθις ε, συζήτηση που κάνουμε σε αυτήν την Επιτροπή. Ορισμένοι από τους συναδέλφους αναφέρθηκαν στα επιχειρήματα ε, της ε, σύντομης επεξήγησης. Άλλοι παρέκλειναν πολύ από το πεδίο της γνωμοδότησης και για κάποιους θα μπορούσα να πω ή θεωρούν ότι υπάρχει κακόπιστη προσέγγιση ε, στην γνωμοδότησή μου. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι ευθύς εξ αρχής. Δεν είναι μια γνωμοδότηση υπέρ του προστατευτισμού. Καμία σχέση. Είναι μια γνωμοδότηση που εφιστά την προσοχή στις πραγματικές αρνητικές συνέπειες αυτού του τύπου φιλελευθερωποίησης που τώρα επικρατεί. Και είμαι πεπισμένος ότι αυτή ακριβώς η Επιτροπή είναι αυτή που θα πρέπει όσο πιο σοβαρά μπορεί και υπεύθυνα να τονίσει αυτές τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις αυτού του είδους της απελευθέρωσης ή φιλελευθερωποίησης. Ε, ορισμένοι συνάδελφοι απευθύνθηκαν ε, ε, σε μένα προσωπικά, αν εγώ πιστεύω κτλ, κτλ. Μπορώ να πω ότι και με την προηγούμενη ιδιότητά μου στη Βουλγαρία, εγώ πραγματικά ε, εργάστηκα σκληρά για να ε, ενταχθεί η Βουλγαρία στον ΠΟΕ και γενικότερα ήθελα να συμμετάσχει η Βουλγαρία στο διεθνές εμπορικό σύστημα. Όμως, έχω και την εμπειρία των ε, πολύ σημαντικών ε, αρνητικών συνεπειών ε, που εντοπίστηκαν στη Βουλγαρία. Και εξετάζοντας και την κατάσταση στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, δεν χρειάζεται να πω στον κόσμο να, να εξετάσει μελέτες, είτε έχουν αξιολογηθεί από ομοτήμου είτε όχι, για να κατανοήσουν την κατάσταση. Αναφέρθηκε το θέμα των μοντέλων. Η κυρία Χάρκιν πολύ σωστά ανέφερε Ε, την πραγματικότητα αυτών των στατικών μοντέλων που αγνοούν το μικρό αυτό ότι υπάρχει ανεργία στον κόσμο, ότι δεν υπάρχει πλήρης απασχόληση στον κόσμο. Και αυτό είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, αλλά και η Βόρεια Αμερική. Ας είμαστε σαφείς λοιπόν. Εδώ πρόκειται για την γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης που ε, θα δώσουμε στην ε, καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου που τελικά, λαμβάνοντα υπόψη και τι άλλε νομοδοτήσει των άλλων επιτροπών, θα διαμορφώσουν μια ισορροπημένη γνώμη. Όμω, πιστεύω πραγματικά ότι θα πρέπει να ε, αρνητικά η Επιτροπή μα εδώ, για να υπάρχει πλήρη επίγνωση ότι δεν μπορούμε απλώ να κινηθούμε με γενικέ διακηρύξει ότι ε, η πρόταση κινείται προς το γενικό συμφέρον, ε, θα ε, προάγει την δημόσια ευημερία κτλ. Αυτά δεν τα έχω επινοήσει εγώ τα επιχειρήματα. Υπάρχουν σε ευρέως γνωστές μελέτες που θέτω υπό εξέταση όλων των εισηγητών. Μπορείτε να τις αγνοήσετε αν θέλετε ή να αμφισβητήσετε τα στοιχεία. Αλλά δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Μόνο τέτοιες δηλώσεις άκουσα. Και πάλι, αυτό που είπε η Μαρία Αρένα. Προς τι όλη αυτή η βιασύνη για την τελική αξιολόγηση. Γιατί δεν υπάρχει μια περίοδος ε, που να περιμένουμε τη νέα αξιολόγηση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι αυτή του 2011 για να απαντήσουμε υπεύθυνα όλα τα ερωτήματα που ανακύπτουν και όλες τις διαμαρτυρίες. Ε, δεν μας ενδιαφέρει το τι λένε οι πολίτες. Και πραγματικά να περασπιστούμε με έναν πιστικό και ε, συστηματικό τρόπο την πρότασή μας. Όχι, οι συνάδελφοι προτείνουν το αντίθετο. Εγώ παραθέτω, κλείνοντα αυτή την αξιολόγηση αντικτύπου του 2011, που είναι πραγματικά απεσιόδοξη συνολικά κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχουν ε, κάποιες θετικές και πιθανόν κάποιες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ε, την προώθηση των επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη ε, και τα κοινωνικά και εργασιακά ενδέχεται να αυξηθούν και οι κοινωνικές ανισότητες παρότι μπορεί να ε, διαμορφώσει και κάποια ανισότητα στους μισθούς κτλ. Λυπάμαι, αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα για την υποστήριξη της συμφωνίας ΣΕΤΑ. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας. Όλοι γνωρίζουμε το χρονοδιάγραμμα που ακολουθείτε για αυτή την έκθεση. Έχει αλλάξει πολλές φορές η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στην Καθήλυνη Μόδια Επιτροπή ΙΝΤΑ θα ψηφιστεί στις 22 Ιανουαρίου. Έχει αλλάξει η ημερομηνία και στην Ολομέλεια θα περάσει στη συνέχεια. Σε 9 λεπτά θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της ε, πρωινής μας ε, συνεδρίασης και ελπίζω όσοι συμμετείχαν ε, στη συζήτηση για τη ΣΕΤΑ να μείνουν. Γιατί θα έρθει η Επίτροπος ε, Μάλστρομ και θα έχουμε και τον πρόεδρο της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ, τον κύριο Μπέντ Λάγκε. Ένα λεπτό διάλειμμα λοιπόν και συνεχίζουμε. Thank you uh, for